Okay, good afternoon, Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε λοιπόν την εργασία μας με την απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι χρόνος ψηφοφορίας. Ε, το θέμα της ψηφοφορίας είναι μια γνωμοδότηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας. Ε, έχει εκπονηθεί από την κυρία Νταντσίλα η γνωμοδότηση. Θέλετε να λάβετε το λόγο, να μας πείτε μερικά λόγια πριν ψηφίσουμε. Όχι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σας θυμίζω ότι θα πρέπει να είστε έτοιμοι με τις κάρτες για να ψηφίσετε, γιατί καμιά φορά χρειάζεται να εξακριβώσουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Για την ενημέρωσή σας είχαμε πάρα πολλούς, πολλές τροπολογίες, 22 συμβιβασμούς και θα ακολουθήσουμε το σχέδιο καταλόγου ψηφοφορίας που έχετε ενώπιόν σας. Αρχίζουμε με την τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Σε αυτή την περίπτωση περνάμε στην τροπολογία 79 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 8. Έχουμε μια, ένα αίτημα προφορικό της ε, εισηγήτριας, όχι. Πολύ καλά. Βλέπετε λοιπόν το κείμενο της ε, προφορικής τροπολογίας. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 22, συμβιβασμός 22. Υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 83 υπέρ κατά άποχες δεκτή. Συμβιβασμός υπαριθμών 1 υπέρ κατά άποχες δεκτή, δεκτός. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια δεν θέλει να λάβει τον λόγο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Συμβιβασμός 4. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτός. Τροπολογία 92. Προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, δεκτό. Συμβιβασμός 5. Υπέρ, κατά, αποχές, Δεκτός. Τροπολογία 15. 16 μάλλον. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβασμός 6. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 97. Υπέρ, 97 υπέρ, κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 97 και θα ζητήσω να αρχίσουμε τώρα την ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. «21 υπέρ, 14 κατά και 2 αποχές». Συνεπώς, η τροπολογία εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τώρα με την τροπολογία 98, καταπίπτει Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα συμβιβασμός 8. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 23 ε, υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Ε, προφορική ε, τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στον συμβιβασμό 11. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 13. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία... Όχι, όχι, λάθος, ναι. Τροπολογία 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 123. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 124. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτε. Όχι, όχι, εγκρίνεται, με συγχωρείτε. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 127. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να πείτε τίποτα εφόσον υπάρχει προφορική τροπολογία, όχι. Απολογία 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ

αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, να κάνουμε θέση. Τροπολογία 37. Ψηφίζουμε την τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, 20 κατά. Ε, απορρίπτεται λοιπόν. Περνάμε στην τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 με προφορικό αίτημα από την εισηγήτρια. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε το προφορικά αίτημα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 148. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να κάνουμε παλήθευση. Τροπολογία 148, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα με την ψηφοφορία. Υπάρχει ένας επιπλέον ε, από το ΕΛΚ. Ωραία, επομένως πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 148. Πέραση της ψηφοφορίας. 16 ψήφοι υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 152. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Τροπολογία 152. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκαεννέα ψήφοι υπέρ. 16 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται η τροπολογία. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 45. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48 με προφορικό αίτημα της ε, εισηγήτριας. Θέλετε το λόγο. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν το προφορικό αίτημα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τώρα. Με την τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 50, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 18 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Πρέπει να περάσουμε πρώτα από την τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 64, προφορικό αίτημα, δεν θέλετε το λόγο. Ψηφίσουμε λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 69. Προφορικό αίτημα. Δεν θέλετε το λόγο. Ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τώρα. Συμβιβαστική τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 73, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 με προφορικό αίτημα της συντάκτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία γιατί εγκρίθηκε η τροπολογία. Επομένως ψηφίζουμε ηλεκτρονικά να ξεκινήσουμε άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 37 ψηφίσαντες, 29 υπέρ, 6 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ την συντάκτρια της νομοδότησης και ευχαριστώ και την Επιτροπή. It was, it was a good job. Τα πήγαμε καλά με την ψηφοφορία. Να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Τον Ιούλιο του 2014 η Επιτροπή υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης ώστε οι μικροπιστές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας. Αφορά πολλές πτυχές ε, πράσινης ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις και για την ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων και τη δημιουργία μιας αλυσίδας αξιών. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης αποφάσισε να ευθύσει μια γνωμοδότηση γιατί ο ε, ε, περιορισμό των εκπομπών ε, είναι κάτι που Ο εισηγητής είναι ο κύριος Νίκα, ο οποίος δεν παραβρίσκεται εδώ σήμερα. Η πρότασή μου είναι η εξή. Έχουμε το σχέδιο έκθεσης από τον εισηγητή μπορούμε να δώσουμε μια προθεσμία για υποβολή τροπολογιών για την 5η 5 Μαρτίου και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε προς το παρόν να κλείσουμε αυτό το θέμα από την ημερήσια διάταξη και να παραλάβουμε απευθείας τις ε, τροπολογίες ε, στην καταληκτική προθεσμία. Συμφωνείτε, συμφωνούν και οι σκιώδεις συγκητές. Σας ευχαριστώ. Σας πενθυμίζω, 12 η ώρα το μεσημέρι, 5η 5 Μαρτίου είναι προθεσμία για υποβολή τροπολογιών για την σχέδιο γνωμοδότηση σχετικά με τις κυρίες πράσινης ανάπτυξης της και μεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε στο επόμενο σημείο της μέρης διάταξης. Thank you for shutting mouths. <laughs> Okay, the next point in our agenda is uh, European Fund for Strategic. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Βανίστερ Λόι. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί δέχτηκε να προετοιμάσει αυτή την έκθεση σε πολύ ε, πιεστική προθεσμία. Η έκθεση παρουσιάζεται στα μέλη της Επιτροπής στα αγγλικά. Τους παρουσιάστηκε λοιπόν και σήμερα θα συζητήσουμε σχετικά με αυτή τη γνωμοδότηση και θα ψηφίσουμε στη συνεδρίαση του Μαρτίου. Η καταληκτική προθεσμία για υποβολή τροπολογιών που προτείνω είναι μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, 5η. Μόνο στα αγγλικά παρακαλώ οι προτάσεις και οι τροπολογίες. Είμαστε πιεσμένοι χρονικά με αυτή την έκθεση, σας το υπενθυμίζω, ε, είναι δύσκολες συνθήκες. Έχουμε επομένως ε, την έκθεση στα αγγλικά και θέλουμε και οι τροπολογίες ε, να είναι στα αγγλικά υποβολή μέχρι 5 Μαρτίου. Άλλο τρόπο για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Ο κύριο Βανίστη Λρόι δέχτηκε να είναι εισηγητή για το επόμενο σημείο τη ε, ημερησία διάταξης. Σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού αριθμό 1 19-15 Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Καθώ οι δύο εκθέσει σχετίζονται θα μας ενημερώσει και για τις δύο ταυτόχρονα. Συμφωνείτε κύριε, Βαν, ε, Ρόι. Είστε σύμφωνος με αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ο λόγος εσάς κύριε ε, Ρόι. Θα μιλήσω αγγλικά. Καθώς επιτρέπετε μόνο στα αγγλικά να εργαζόμαστε, πότε κατάλαβα. Στην διπλανή αίθουσα Υπάρχει μια διαδικασία ερωταποντήσεων για τους εισηγητές. Λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να είμαι στο 4Q, 4Q1. Ε, Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε διπλές ε, υποχρεώσεις. Στην πράσινη εβδομάδα κάποιοι εργάστηκαν σκληρά για να έχουμε ένα ισορροπημένο έγγραφο και να ε, παραμείνουμε στις αρμοδιότητες και στις ευθύνες της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπάρχει μεγάλη ένταση στις Επιτροπές ε, Ίντερα και στην Επιτροπή Μεταφορών. Ο δικός μας ο δεν αγγίζεται άμεσα γιατί έχουμε δύο τελείως διαφορετικά ε, εργαλεία και είναι πολύ σημαντικό το Ταμείο Συνοχής να μην συνεισφέρουν άμεσα στο Ταμείο Εγγύησεων, το Ταμείο Επενδύσεων ε, του Γιούγκερ. Αυτό είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε ώστε να ελέγξουμε τα που θα γίνουν προς τα κάτω, ώστε να χτίσουμε και συνέργειες. Με αυτόν τον τρόπο το εξέτασα το θέμα. Το νέο ταμείο θα συνεισφέρει στους ε, στόχους για την κοινωνική και ταφική συνοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο το εξέτασα και έτσι λοιπόν δεν έψα στην παγίδα γιατί υπάρχουν και άλλες επιτροπές με εκτεταμένες υποχρεώσεις κτλ. Οπότε καλό είναι να παραμείνουμε στις αρμοδιότητες μας και στις ευθύνες μας ως ε, επιτροπή. Κρατά το έργο μας ε, ζωντανό. Το νέο ταμείο λοιπόν, όπως είπα, δεν θα πρέπει να κανιβαλίσει Ε, στα επενδυτικά ταμεία. Γιατί αν μπορούμε να λάβουμε με εύκολο τρόπο χρήματα, θα έρθουν πολλοί από την Τράπεζα Επενδύσεων στη Ρουμανία και θα πούν «Ναι, θα σας βοηθήσουμε να πάρτε τα κονδύλια και αυτό θα τους ε, δημιουργήσει σύγχυση. Και μπορεί κάποιοι να να επιλέξουν το νέο ταμείο γιατί θα πληρώσει ενδεχομένω καλύτερο. Λοιπόν, προσοχή. Μπορούμε να κάνουμε κασίες. Δεν ξέρουμε όμω στην πράξη πώ θα λειτουργήσει αυτό. Στην παρούσα κατάσταση υπάρχει μια θετική προσέγγιση. Και κατά δεύτερον, ναι, θα έχουμε συνέργειε στις χώρες όπου γίνονται προγράμματα υποδομών, έρευνα κτλ. πληροδικά προγράμματα στον τομέα τη ενέργεια, παραδείγματο χάρη. Και που σε κάποια φάση ε, ε, που ήδη χρηματοδοτούνται από κάποια από τα ταμεία. Στην περίπτωση που θα ολοκληρωθούν αυτά τα προγράμματα. Και με την παροχή εγγύσεων από τα νέα ταμεία. Αυτά μπορούν να συμβούν και είμαι πολύ θετικά διακείμενος γιατί μπορεί να προχωρήσει αυτό. Και τα διευθυντικά επενδυτικά ταμεία δεν αποκλείουν τέτοιου είδους δραστηριότητες κατά δεύτερον. Το νέο ταμείο παρέχει τη δυνατότητα για πλατφόρμες ανανέωσης στις ε, χώρες και στις περιφέρειες. εντάσσονται και άλλα χρηματοδοτικά μέσα και βλέπω ότι οι αρχές οι οποίες αναλαμβάνουν τα έργα είναι οι ίδιες ομάδες ανθρώπων με αυτές που προετοιμάζουν πρωτοβουλίες για τα διευθυντικά ταμεία. Και γι' αυτό στις τροπολογίες Έχω δύο σημαντικά, έχω δύο σημαντικά στοιχεία. Κάνω αναφορά στις προτεραιότητες των περιφερειακών ταμείων επενδύσεων και τονίσω την δυνατότητα να υπάρξουν συνέργειες. Επιπλέον θα ήθελα να πληροφορηθώ για τον αντίκτυπο που θα έχουν τα νέα, το αντίκτυπο που θα έχει το νέο ε, ταμείο. Αυτό είναι ένα στήμα αξιολόγηση. Γιατί μπορεί το ταμείο να λειτουργήσει θετικά σε σχέση με την οικονομική χρήση, κρίση. Π.χ. στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία όπου υπάρχει μεγάλη διαρροή νέων. Αυτό το νέο Ταμείο να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Ε, να έχει θετικά αποτελέσματα για τις ε, Μητροπόλεις και να επιδράσει αρνητικά στην ε, Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές. Άρα χρειάζεται να γίνει μια αξιολόγηση. Πρέπει να έχουμε επομένως αυτή την ενημέρωση, αυτή την αξιολόγηση. Γιατί για μισή ώρα άκουγα δίπλα ότι πρέπει να έχουμε βιώσιμα έργα. Αλλά μισό λεπτό, ε. υπάρχουν ε, περισσότερα θέματα εδώ. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε εκ των προτέρων αυτή την ε, αξιολόγηση. Και περαιτέρω, επιπλέον, εισήγαγα κάποια σημεία σε σχέση με το τι σκοπεύουμε να κάνουμε για τις ε, ανισορροπίες, για τη διασυνοριακή διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό μεταξύ χωρών να ληφθούν υπόψη αυτές οι διαστορεικές ε, πτυχές. Και μέσα στα έγγραφα βλέπουμε τον επιπλέον συμπληρωματικό χαρακτήρα αυτού του νέου ταμείου. Γιατί ε, τα δημόσια χρέη που υπάρχουν, αν χρηματοδοτηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε δεν υπάρχει προστιθέμενη ποιότητα και αξία. Αν όμως ε, πράγματι συμβεί αυτό, δεν υπάρχει ουσιαστική κοινωνική ε, συνεισφορά. Άρα θέλουμε να έχουμε επιπρόσθετη, επιπρόσθετες συνεισφορές και όχι αντικατάσταση. Μια τελευταία παρατήρηση για το σημείο αυτό της σημερινής διάταξης. έχει να κάνει με τα γεωγραφικά κριτήρια. Είναι κάτι που δεν το θεωρώ απαραίτητο, γιατί γεωγραφικό σημαίνει ότι, ε, ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε θα πρέπει να ε, έχει πρόσβαση σε αυτά τα κονδυλία Γαλλία, Ιταλία, παραδείγματο χάρη. Μένω λοιπόν σε ένα πιο γενικό επίπεδο και προσπαθώ ε, να υπάρχει μια ισορροπία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η συνεισφορά που θα υπάρχει για την ε, κοινωνική, οικονομική και ε, δαφική συνοχή. Και να περάσουμε και στην, ε, στο επόμενο σημείο για την αναθεώρηση του προπολογισμού. Διότι το, δεν θα πρέπει το Ταμείο να έχει αρνητικές επιστώσεις, επιπτώσεις πάνω στα όσα υπάρχουν. Θα πρέπει να είναι το νέο Ταμείο να έχει 1,5 χρόνο και να υπάρχει μια προσέγγιση ε, βιώσιμη, διαρθρωτική και πάλι να μπορέσουν ε, να συμμετάσχουν με χρήματα στο επίπεδο των έργων. Ούτως ώστε τα έργα αυτά, τα προγράμματα αυτά, βάσει του νέου ε, ταμείου, να αποδώσουν όχι μόνο στο, όχι στο επίπεδο του ίδιου του προϋπολογισμού, αυτή είναι η παρέμβαση που ήθελα να κάνω και είμαι στη διάθεσή σας και μπορώ να δεχθώ τροπολογίες. Είναι τα γενέθλιά μου, είτε μου φέρετε ένα γλυκό, είτε μία τροπολογία. Τα είναι project. Thank you very much for this very Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρέμβαση και προσέγγιση της έκθεσης. Θα έχουμε το Μάρτιο, στη συνέχεια. είναι ο σκιώδης εισηγητής. Η κυρία Μπρέσο έχει το λόγο. Italian. I know that... Ναι, μπορώ να μιλήσω Ιταλικά. Ξέρω ότι πρέπει να γράψω στα αγγλικά, αλλά πρέπει να μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστώ. Επειδή πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι μάλλον περίπλοκο, προτιμώ να τα πω στη γλώσσα μου. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να τον διαβεβαιώσω ότι θα λάβει τροπολογίες από εμά. Θα ξεκινούν με χρόνια πολλά και μετά από εκεί και πέρα θα σας ε, υποβάλω τις υπόλοιπε ε, τροπολογίες. Απλώς για να μην ξεχάσουμε και τα γενέθλιά σας στις 5 Μαρτίου. Η γνωμοδότηση και οι τροπολογίες που μας παρουσίασε ήδη είναι ενδιαφέρουσες και από μια γρήγορη ματιά που ρίξαμε, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε και συμφωνούμε και με την ανάλυση που μας παρουσιάζεται. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και βεβαίως από εκεί και πέρα θα αξιολογήσουμε ποιες ε, τροπολογίες θα σας καταθέσουμε. Η πρώτη μου παρατήρηση, η οποία ε, είναι προς την κατεύθυνση αυτών που μας είπατε είναι ότι αυτό το ε, ταμείο προσφέρει εγγυήσεις, όχι επιπλέον χρήματα, διότι ούτως ή άλλως θα ε, έπρεπε να τα βρούμε από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα πάντα έχουν διατεθεί. Επομένως ήταν δύσκολο. Θέλουμε να προσερκίσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και κυρίως ε, θεσμικούς επενδυτές για να μπορέσουμε να δώσουμε νέα όθεση στις επενδύσεις. Επενδύσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι επενδύσεις οι οποίες θα είναι σε θέση να οδηγήσουν σε απασχόληση και ε, σε εισοδήματα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ε, αυτή της μορφή επενδύσεις ε, θα πρέπει περισσότερο να τίνουν στον εξυγχρονισμό του παραγωγικού μας ιστού ή του συστήματος υποδεμών και διασυνδέσεων και όχι ε, για να αυξήσουμε την παραγωγική μας ικανότητα που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι μάλλον υπερβολική ήδη. Ε, μάλλον θέλουμε να συγχρονίσουμε τα πράγματα και να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα καλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενώπιον του, ε, για τις υποδομές μας συγγνώμη, και για το παραγωγικό μας σύστημα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πραγματική προστιθέμενη αξία. Επειδή ε, στην ουσία εδώ αναφερόμαστε σε εγγυήσει, σε πολλές περιπτώσεις, εάν οι επενδύσεις μπορούν να συνδεθούν έχοντας ταυτόχρονα και χρηματοδότηση για το από το ιδιωτικό σύστημα χρηματοδότησης δεν θα υπήρχε λόγος ε, για εγγύσεις. Το θέμα λοιπόν της προστιθέμενης αξίας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στόχος μας πρέπει να είναι να αυξήσουμε την ποσότητα των επενδύσεων και όχι να υποκαταστήσουμε μια δημόσια εγγύηση ε, με μια ιδιωτική εγγύηση. Και από αυτή τη σκοπιά δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι η συνέργεια με τα διαρθρωτικά ταμεία που πολλές φορές υπενθυμίζεται από τον ε, ε, συντάκτη της νομοδότησης είναι πάρα πολύ σημαντική διότι το σύστημα για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες είναι νέο και επομένως είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω επενδύσεις, ιδίως όταν απευθύνεται ε, στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να συνδυάζεται και με τις ε, υφιστάμενες επενδυτικές προσπάθειες, ε, τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχει μεικτή χρηματοδότηση και από δημόσια και από ιδιωτικά κονδύλια. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ε, ωστόσο, οι επενδύσεις του σχεδίου Juncker να υποκαταστήσουν τρόπον τεινά τις επενδύσεις των διαρθρωτικών ταμείων και να τα μεταφέρουν προς δραστηριότητες που δεν είναι και τόσο παραγωγικές από πλευράς απασχόλησης και εισοδήματος. Θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει συνέργεια και πραγματικά να βοηθούν να υπάρχει αποτελεσματικότητα και αποτέλεσμα στα διαρθρωτικά ταμεία. Όχι να τα μετατοπίσουμε προς κάποιες άλλες μορφές επενδύσεων που δεν είναι και πολύ αποτελεσματικές και πολύ παραγωγικές τέλος δεν θα έχουμε αυτό το επιπλέον αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε. Να υπενθυμίσω ότι Σαφώς ε, και ισχύει το θέμα της εδαφικής ισορροπίας. Ο στόχος οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πολιτικής πρέπει να είναι η εδαφική συνοχή. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε επενδύσεις που να αντιβαίνουν στην αρχή της εδαφικής συνοχής. Και επίσης να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν και κάποιες χώρες παρόλα αυτά όπου το 3α ε, ουσιαστικά προσδίδει ελάχιστη ουσία σε ένα ε, σύστημα εγγύησεων. Στην πραγματικότητα οι εγγύησει θα ε, στοχεύουν κυρίως στις επενδύσεις. Σίγουρα ιδιωτικές και επενδύσεις από θεσμικούς επενδυτές, κυρίως εκεί όπου το επίπεδο της αναγνωρισμένης ευρωστίας του κράτους είναι πιο χαμηλό και επομένως υπάρχει κίνδυνος για τις επενδύσεις ε, είναι, και είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος από όπου αλλού. Ε, και αυτός είναι ο στόχος ο οποίος ε, σαφέστατα υποδεικνύεται στο πρόγραμμα. Κάτι επιπλέον. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς κινούμεθα προς τη μεγαλύτερη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων, θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποιος συντονισμός και μία απλούστευση ως προς τη χρήση αυτών των μέσων, ακόμα και ε, στα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα διαρθρωτικά κονδύλια. Και κάτι τελευταίο, εάν καταφέρουμε για μεγάλα προγράμματα εδαφικά, τα ε, κονδύλια από το σχέδιο Juncker, ακόμα και υπό τη μορφή επενδύσεων, ουσιαστικά η δημιουργία επενδύσεων με το σχέδιο Juncker, αν μπορούν να έχουν κάποιες συνέργειες με τις επενδύσεις των διαφθορτικών ταμείων, σίγουρα θα αυξήσουν και τις δυνατότητες των διαφθορτικών ταμείων να δώσουν μια νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδίω να την δώσουν στις περιοχές τις οποίες επλήγησαν ε, περισσότερο στη διάρκεια αυτής της κρίσης και που ε, ακόμα έχουν όμως πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Όπως σας έλεγα, ε, προφανώς ε, μέχρι τις 5 Μαρτίου, μαζί με τις ευχές προς τον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης, θα στείλουμε και κάποιες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλοι σκιώδεις εδώ. Ο κύριος Λουέρ. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να μην χάσω το τρένο μου, παρόλα αυτά θέλω να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση βλέπω ε, ότι πρέπει να δούμε πώς θα, στο πρόγραμμα αυτό θα εντάξουμε την συνοχή, διότι θα ήταν κάτι το χρήσιμο. Έχουμε όμως χρήματα από το ορίζον 2020, τουλάχιστον ως προς τις προθέσεις του ε, προγράμματος Juncker και έχουμε ορισμένα προγράμματα, προγράμματα ε, και σχέδια ε, συνοχής ε, σε σχέση με τα χρήματα που θα ξοδευτούν, τα κονδύλια που είναι απλώς για έρευνα. Είναι προϊόντα που θα έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά εξακολουθώ να έχω ανησυχίες και επιφυλάξεις για την αντίληψή του να διαλέγουμε κερδισμένους και ότι δεν πρέπει να ασχολούμεθα με το Horizon 2020 ε, διότι θα καλυφθεί με τις αποδόσεις ε, των επενδύσεων, τα κέρδη των επενδύσεων. Οι ιδιώτες χρηματοδότες ε, κρίνουν τις επενδύσεις αλλά το κράτος ή το υπερκράτος δεν ξέρω τι θα σκεφτεί για τις επενδύσεις, αμφιβάλλω και αμφιβάλλω ότι, αν, ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια ε, θα προσεγγίσουν επίπεδο, το επίπεδο που επιθυμεί ο Γιούγκερ. Τα 350 δισεκατομμύρια. Και ε, δεν μπορώ να συμμεριστώ την ε, αισιοδοξία αυτών των προτάσεων και πρέπει όμως να εξετάσουμε τα πραγματικά αποτελέσματα για να δούμε ε, και την άλλη πλευρά, δηλαδή να δούμε ε, τα, αποτελε... τα αίτια και τα... τις συνέπειες τους. Αν υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν θα πούμε «Α, απλώς είναι μεγάλη επιτυχία το σχέδιο Juncker». Πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές, ε, ρεαλιστικά να σταθμίσουμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαμπό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα και καταρχήν είμαι πολύ ικανοποιημένος που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ στην αίθουσα και όπως έλεγε και ο ε, εισηγητής έρχομαι από τη διπλανή αίθουσα. Εκεί είχαμε μία συνάντηση που συζητούσε ε, για το σχέδιο Juncker. Και θεωρώ ότι δίπλα ή τουλάχιστον έτσι εμένα μου φάνηκε, ότι βρέθηκα κάπου μεταξύ ενός ε, ε, τραπεζικού γραφείου και ε, οικονομικών συμβούλων. Και εγώ είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύω ότι μας εξέλεξαν εμάς όλους για να κάνουμε πολιτική και για να ασχολούμαστε με το λαό. Ε, συζητούσαν το ε, αν θα πρέπει να πάμε από το 13 στο 15 γιατί τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως ότι δεν θα πρέπει να εθνικοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις, διότι όπως έλεγε και ο εισηγητής μας, ούτως ή άλλως ε, τα χρήματα είναι χρήματα και θα πρέπει ε, να προσέξουμε γιατί θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε απλώς τους πλουσίους. Εντάξει, δεν θέλουμε να τα εθνικοποιήσουμε. Αλλά εάν φτάσουμε στα άκρα και πάλι ελοχεύει κάποιο κίνδυνο. Γιατί μπορεί να κάνουμε επενδύσει τελικά στην Ιαπωνία ή στον Delaware. Και δεν νομίζω ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό με το σχέδιο Juncker. Τι εννοώ με αυτά τα αστιάκια. Σοβαρά τώρα. Όλοι εμεί, όχι μόνο ο κ. Juncker, όλοι εμεί Εάν δεν καταφέρουμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα εξάλλου. Όχι ότι το μέλλον θα είναι θηλιακό και θα είναι παράδεισος, αλλά σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα οι επενδύσεις του σχεδίου Juncker να επιταθούν ε, απευθείας στην ανεργία θα αποτελέσει μια κοινωνική αποτυχία που θα πλήξει πάρα πολύ την Ευρώπη. Αυτό είναι διαμφισβήτητο. Δηλαδή, το να μπορέσουμε να έχουμε επενδύσεις οι οποίες θα είναι καρποφόρες θα είναι πάρα πολύ καλό. Εάν ο πληθυσμός όμως των χωρών που έχουν τη περισσότερο, περισσότερο δεν το αντιληφθεί ως μείωση της φτώχειας και της ανεργίας, τότε σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό για όλη την Ευρώπη. Εγώ δεν θέλω να τα ε, περιφερειοποιήσουμε, να τα εθνικοποιήσουμε, τίποτα άλλο. Αλλά... Ε, οι άλλες επιτροπές που δεν είναι απλώς και μόνον ε, λογιστικά και οικονομικά θα πρέπει να καθαρίσουν και το πολιτικό σκέλος αυτού που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Θεωρώ ότι οι περιφέρειες και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, πρέπει να επαγρυπνεί ώστε η επιλογή των επενδύσεων που θα γίνουν να έχει ή τουλάχιστον να έχουν την πρόθεση να έχουν αποτελέσματα στον τομέα της ανεργίας και να πω και κάτι ακόμα. Και στις μεγάλες ε, ε, αγορές της απασχόλησης και θα αναφέρω τώρα μια χώρα που αγαπώ πολύ αλλά το να περάσουμε στο Λουξεμβούργο από το 3,0 στο 2,9% ε, δεν έχει και καμία σημασία θέλουμε τις μεγάλες αγορές απασχόλησης να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και νομίζω ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει πολλά να πει και μπορεί να βοηθήσει διότι οι ε, κυβερνήσεις των περιφερειών είναι πολύ πιο ε, κοντά στα κοινωνικά προβλήματα, στα πραγματικά προβλήματα της ανεργίας, της ανεργίας των νέων από ότι προφανώς ε, τα μελετητικά γραφεία ή τα πιο υψηλά επίπεδα διακυβέρνησης που βρίσκονται πιο μακριά. Επομένως, οι τροπολογίες του υποφαινόμενου με πάσα ταπεινότητα θα προσπαθήσουν ε, ε, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να μην ξεχάσουν την ευαισθησία της πολιτικής βαρύτητας αυτού του σχεδίου Βίνκερ. Και καλό όλους τους υπολείπους, πολλό δε μάλλον τον ίδιο τον εισηγητή, να μην ε, παραγωνίσει σε καμία περίπτωση αυτή την αποστολή καταπολέμησης της ανεργίας για να μπορέσει να αντισταθμίσει την απαραίτητη ανάγκη να είμαστε λογικοί και αυστηροί στην επιλογή. Ε, δεν ε, θέλουμε να κάνουμε φτηνό και ινσιανισμό μικρής διάρκειας. Α, σε αυτό συμφωνώ, αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνουμε και γραφείο ελέγχου του κινδύνου και τίποτα άλλο, μια, μιας τράπεζας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ομαρζέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, διότι έχω κι εγώ ένα τρένο. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, η Επιτροπή μας όντως πρέπει να θέσει ένα ερώτημα το οποίο είναι σημαντικό. Αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μήπως επιδεινώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να οδηγήσει σε υποχώρηση της εδαφικής συνοχής. Αυτή είναι η ερώτηση και ξέρουμε λόγω όλου του σκεπτικού ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα κάνουν προτάσεις για περιφέρειες, όχι τις, ε, τις πλουσιότερες, ε, τις πλουσιότερες, τις πιο ανεπτυγμένες και εκεί όπου η ανεργία είναι η πιο μαζική, εκεί όπου υπάρχει μια πραγματική ε, προσδοκία για επενδύσεις, ε, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ανεργίας, αυτές οι περιφέρειες ίσως βρεθούν αποκλεισμένες. Ε, παίρνω τις υπερπεριφερειακές περιοχές, εκεί όπου έχετε ένα, μια ανεργία ρεκόρ, είναι προφανές ότι με τις σημερινές συνθήκες δεν βλέπω λόγω των όσων ε, εγκρίθηκαν, ποια προγράμματα, ποια έργα θα ε, γίνουν σε αυτές τις περιφέρειες από το Ταμείο. Υπάρχει λοιπόν ένα πραγματικό πρόβλημα που τίθεται, γι' αυτό ο εισηγητής δικαίως ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να στηριχθούμε στην ε, συνθήκη για να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οφείλει, οφείλει ε, να τηρήσει ορισμένους στόχους οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής ε, συνοχής, στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Όσον αφορά τα προβλήματα, τα γεωγραφικά, είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει αυτήν την επιλογή και δεν πρέπει αλλά εμείς δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Εμείς, Περιφερειακή Επιτροπή, έχουμε κάνει επιλογή να κατηγοριοποιήσουμε τις περιφέρειές μας και αν το κάναμε είναι επειδή έχει ένα νόημα οι περιφέρειές μας να καταταγούν ανάλογα ε, με την, ε, τις πιο, την ανάπτυξή τους και νομίζω ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επενδύσει θα επενδύσει στο σύνολο της Ευρώπης θα πρέπει να εμπνευστεί από αυτά τα κριτήρια ε, που εμείς υπερασπιζόμαστε. Αυτό ε, μπορεί η Επιτροπή μας ε, να βοηθήσει να γίνει εφόσον κάθε Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξετάσει από κάποιο άποψη το, το σχέδιο Juncker, δημοσιονομικό, δημοσιονομική άποψη ή άλλη. Ε, συνεπώς δεν μπορούμε να περιμένουμε την ε, εργασία άλλων επιτροπών για να τηρήσουμε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζέλλερ νομίζω ζήτησε ε, τον λόγο εσείς και μετά, και μετά εσείς κύριε Βέρκο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα πρέπει να δυσκολέψουμε τα πράγματα και τη δουλειά μας, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες επιτροπές, αλλά να επικεντρωθούμε σε αυτά που είναι σημαντικά για εμάς. Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και για εμάς είναι σημαντικό ότι υπάρχει μία περίοδος παράτησης όπου υπάρχει πολιτική συνοχή, όπου αποκινούμε τα κράτη-μέλη και τις ε, και με την βοήθεια των ε, ταμείων και με τη χρηματοδότηση Τίθενται σε εφαρμογή έργα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Αυτά συζητάμε το... σήμερα σχέση με το, με το σχέδιο Juncker το οποίο έχει μία άλλη ε, επιδίωξη να δημιουργήσει ανάπτυξη στην Ευρώπη και λόγω της δυσκολής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε που εν μέρη έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη σε κάποια αλλά από την άλλη πλευρά ε, σε ιδιωτικά ταμεία υπάρχουν ε, πολλά χρήματα Το σχέδιο του Πρόεδρου της Επιτροπής είναι να δοθεί μια ευκαιρία να δημιουργηθούν επενδύσεις χωρίς να είναι υψηλό το ρίσκο για, τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έτσι το ερμηνεύω εγώ αυτό. Επομένως, ε, έχει να κάνει με το τι θέλουμε εμείς σε σχέση με την ε, ε, πολιτική συνοχής. Και γι' αυτό τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να ε, έχουν ως σκοπό τη μείωση, την λεκτοποίηση του κινδύνου παράλληλα με μια συγχρονοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και έτσι, με αυτή την ικανότητα μόχλευσης, θα είμαστε ικανοί έργα που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι στιγμής να λάβουν χρηματοδότηση. Θα διτεθούν κονδύλια στο πλαίσιο του προπολογισμού από τη μία στην τίμη την ε, έρευνα και την ε, καινοτομία και από την άλλη στον τομέα των μεταφορών. Δεν θα πρέπει να αγγίξουμε τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται για την ε, πολιτική συνοχή. Υπάρχουν όμως κάποιοι που λένε γιατί αντλούμε χρήματα από τον τομέα της έρευνας και από το Connecting Europe Facility και το 2020 Και γιατί δεν παίρνουμε, δεν αντιλούμε κονδύλια από, ε, από θέματα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι ε, στιγμής ε, για τα διευθυντικά ταμεία ή για την ε, γεωργία. Και εδώ θέλω να πω ότι κάτι δεν θα πρέπει να συμβεί. Γιατί θα πρέπει να θυσιάσουμε την περιφερειακή πολιτική και την ε, πολιτική συνοχής ε, για κάτι άλλο. Θα πρέπει να σπάσει το κεφάλι Επιτροπή Προϋπολογισμού αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από το ορίζοντα 2020, από το Connecting Europe Facility κτλ. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς να μην ε, υπονομευθεί η πολιτική συνοχή και τα κονδύλια που προβλέπονται για αυτήν. Και να μην εφαρμοστούν, να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκόπους όπως ένα σχέδιο επένδυσης. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο να συνεχίσουμε την ε, πολιτική συνοχής ε, με το 2020 όπως το έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ, κυρία Ρέιντκε. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της αδελφού ε, Βάνερου που είναι σιώδη ε, εισηγήτρια και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα γιατί πρέπει να επιστρέψει στη Βιέννη. Θα μιλήσω γερμανικά γιατί έχει γράψει τις σημειώσεις της στα γερμανικά να ευχαριστήσω την Γραμματεία και τον εισηγητή που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να εργαστεί τόσο επιτυχώς. Είναι πολύ ε, ε, εύστοχη η έκθεση σε σχέση με το ε, Ευρωπαϊκό Διευθυντικό Ταμείο και σε κάποια σημαντικά σημεία. Η Επιτροπή Περιφερικής Ανάπτυξης με τόσο μεγάλη ε, εμπειρία στην πολιτική συνοχή, είναι σημαντικό να προωθήσει θέματα που αφορούν την απασχόληση και να μην ε, εκτοπιστούν θέματα που αφορούν ε, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρου στόχου για τη δημιουργία θέσεων εργασία σε περιφέρειε με υψηλά ποσοστά ανεργία και να υπάρχουν και συνδευτικά μέτρα για επενδύσει στην εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάσουμε στη δημιουργία θέσεων ε, ε, εργασίας, δικαιωμένων θέσεων εργασίας. Με το Διευθυντικό Ταμείο έχουμε ένα εργαλείο ώστε η επένδυση να έχει ξεκάθαρα κριτήρια ως προς τους στόχους ε, για την Ευρώπη 2020. Θα πρέπει υποθετικά να εμπλακούν οι τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών. Αυτές οι προδιαγραφές όμως λείπουν από το ε, Επενδύσεων. Υπάρχει έλλειψη στον τομέα στρατηγικών επιδείξεων όχι σε κονδύλια αλλά σε ιδέες. Θα θέλαμε λοιπόν να εργαστούμε τι επόμενε εβδομάδε, ε, επί αυτού του θέματος να οδηγήσουμε στη σωστή κατεύθυνση το πρόγραμμα επενδύσεων γιατί ένα σχέδιο χωρί στόχους και χωρίς δημοκρατικά, ε, δημοκρατικές βάσεις δεν μας ε, ε, βοηθάει να προοδεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταμάτο. Ναι, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον συνάδελφο για την γνωμοδότησή του και να πω ότι συμφωνώ τα όσα θέλουν να έχουμε κάποια πρόσθετα στοιχεία μεταξύ Ταμείο συνοχή και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σίγουρα δεν είναι ταυτόσημα γιατί οι 11 θεματικέ ενότητε του 2014-2020 θέλουν να ενισχύσουν και την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να πούμε όμω το ίδιο για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και πραγματικά εγώ τελώ υποσύγχυση για την υποτιθέμενη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο μέσων. Διότι ω συνήθω αναχεύει ο κίνδυνο μια. Ε, Απόκληση ε, κονδυλίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ε, αντί του Ταμείου συνοχή ε, για το Στρατηγικό Ταμείο. Στην, ε, ε, στο άρθρο 5 παράγραφος 4 λέγεται ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική συνοχή για να συνεισφέρουν στην πολιτική επιλέξιμων προγραμμάτων όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Εγγύησης. Ο συνάδελφος προτείνει κάποιες εγγυήσεις όπως για, ε, κάποιες τροπολογίες παραδείγματος χάρη τη 10 την οποία σας παραδέτω και λέει τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να συνεισφέρουν σε επιλέξιμα προγράμματα στα οποία συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με βάση του στόχου, τι αρχέ και του κανόνε του πλαισίου που ισχύει για το Ταμείο αυτό με συμφωνίε εταιρική σχέση και συγκεκριμένα προγράμματα. Το πρόβλημα δεν έγκυται τόσο στι τροπολογίε του συναδέλφου, διότι είδα και σε άλλα σημεία του κειμένου αναφέρεται στην ανάγκη να λάβουμε υπόψη και του στόχου τη κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τι περαιτέρω ανισότητε στην περιοχή, αλλά στην ίδια την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια τη δική μα τη πολιτική συνοχή για το Ταμείο Στρατηγών Επενδύσεων. Και μάλιστα του δόθηκε η δυνατότητα αυτού του ταμείου να μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, κρατική χρηματοδότηση, να ε, παραβιάσει τους κανόνες για το έλλειμμα, ενώ ε, στο Ταμείο Συνοχής ε, καταλαβαίνετε ότι τα κράτη-μέλη ε, δεν μπορούν να παρεκκλίνουν και μπορεί να υπάρχει βέλη να χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν το στρατηγικό ταμείο ακριβώ για να παρεκκλίνουν από του κανόνε. Κατά την άποψή μου αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επίσης θεωρώ ότι παρά τις τροπολογίες που θα μπορούσαμε να προτείνουμε ώστε να είναι όλο πιο ήπιο το Ταμείο Στρατηγών Επενδύσεων για την ε, Περιφερειακή Πολιτική, αν δεν αντιμετωπίσουμε το βασικό θέμα της ε, πιθανής ε, παρεκτροπής των κονδυλίων, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτα. Όσον αφορά το θέμα της διακυβέρνησης του στρατηγικού αυτού ταμείου, κυρίως όσον αφορά τα μεμονωμένα προγράμματα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο παράδειγμα διαφάνειας και συμμετοχής, διότι φαίνεται ότι θα υπάρχουν έξι εμπειρογνώμονες, εμπειρογνώμονες εμπειρογνώμονες γνώστες στις αγορές, ανεξάρτητοι και θα αποτελείται και από έναν ε, ε, σύμβουλο όλα κατόπιν προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το κοινοβούλιο που είναι. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Novak. Ευχαριστώ κύριος Νοβάκο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε παρόλο που δεν υπάρχει γραπτός κανόνας για γεωγραφικός ε, για τα έργα στην Ευρώπη, ήδη έχουμε μερικές ανισορροπίες στις περισσότερες χώρες. Μερικές περιφέρειες είναι καλά ανεπτυγμένες, άλλες δεν είναι και δεν ε, χρειαζόμαστε άλλο ένα μέσο για να αυξήσουμε τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Ε, θα πρέπει να τονίσω ότι όχι μόνο πρέπει να αποφύγουμε αυτό στην πολιτική συνοχή στο σχέδιο Juncker, αλλά επιπλέον θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργειες ανάμεσα στα δύο αυτά εργαλεία, στα δύο αυτά μέσα, ούτω ώστε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα περισσότερα έργα και προγράμματα και να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία, διότι αυτό είναι που περιμένουν ε, οι λαοί από μας. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν κριτήρια διαφανή για το πώς τα έργα και τα προγράμματα θα γίνουν δεκτά και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει ίση πρόσβαση στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων για να αποφύγει ε, επιφυλάξεις ε, για το ότι μερικές χώρες έχουν περισσότερη επίδραση και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση της ευαισθητοποίησης για το τι κάνει το πρόγραμμα. Υπάρχουν χώρες που έχουν υποβάλει έργα, έργα υδραυλικά δεν ξέρω εάν οι επενδυτές ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους προγράμματα. Θέλουν δημιουργική οικονομία, ε, high-tech, ε, τεχνολογία πληροφοριών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Πρέπει να διευκρινίσουμε ποιος είναι ο βασικός στόχος του σχεδίου Juncker. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει τον λόγο. Κύριε Βαν Λίστερνόη, θέλετε ε, να ε, αντιδράσετε σε ορισμένα από τα σχόλια που έχουν γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στο κείμενό μας έχουμε τα βασικά ε, σημεία αν υπάρχουν μερικά πρόσθετα σημεία στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας είμαι ανοιχτός, αλλά νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα όπως η διακυβέρνηση κλπ. θα συζητηθούν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ας μην προχωρήσουμε πολύ μακριά. Είναι ε, σωστά τα όσα λέχθηκαν. Είναι ε, τελείως άλλη, άλλη άλλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για χρήματα. Πώς ε, είναι ο πολλαπλασιαστής, θα το χάρη, ε, στο ορίζον 1, 15, τι προέρχεται αν βάλουμε ε, τόσα ευρώ, πώς πολλαπλασιάζονται, πώς είναι ο πολλαπλασιαστής. Ο πολλαπλασιαστής δεν είναι τόσο σημαντικός καμιά φορά διότι αρχίζεται στην αρχή να δημιουργείται κέντρα εκπαιδευτικά. Ο πολλαπλασιαστής είναι δύσκολο να βρεθεί τότε διότι πληρώνεται, έχετε έξοδα, έχετε χορηγήσεις, ε, και μερικοί λένε έχετε και υποτροφίες και λένε πολύ ότι αυτό είναι πεταμένο χρήμα, αλλά δημιουργούμε με τα χρήμα. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε την γραμμή που λέχθηκε σε όλη τη συζήτηση να πούμε ότι είναι διαφορετική στόχη, διαφορετικό χρήμα, διαφορετική θέση και που μπορείτε να ευθυγραμμιστείτε, που μπορεί να επενδύσετε, έχετε μια κατάσταση στη χώρα σας, μπορείτε ναι, στη κάθε χώρα ε, να ε, ασχοληθείτε με το θέμα αυτό, αλλά είναι άλλη δουλειά. Πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά αναπτύσσονται γι' αυτό. Θέλω να έχουμε αυτή την αξιολόγηση σε ένα, δύο, τρία χρόνια, περίοδη αξιολόγησης όπου θα εξηγήσουμε ότι οι χώρες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες των όσων κάνουν, διότι τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά στην Ιταλία, στη Σουηδία, πώς γίνεται ο συνδυασμός και τότε θα μπορούμε να έχουμε μια άλλη συζήτηση ενδελεχέστερη για το τι είναι βιώσιμο, τι δεν είναι. Διότι δεν ξέρω, θα υπάρξει ένα είδος, ε, ένας τομέας όπου έχουμε κάποια σύνδεση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ξοδεύουν πεταμένα χρήματα, ε, διότι έχουμε αυτήν την μόχλευση. Υπάρχουν αρκετά χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, που δίδονται χωρίς ε, απόδοση. Το πραγματικό πρόβλημα είναι να υπάρξουν εξελίξεις στις περιφέρειες και στις περιοχές όπου έχετε αυτά τα θεμελιώδη, τα βασικά προβλήματα. Αυτό δεν γίνεται με υψηλέ εγγύησει χρημάτων. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, θα επικοινωνήσουμε. Δεν είμαστε αρνητικοί ω προς το Ταμείο Juncker καθόλου, αλλά θα πρέπει ε, να δημοσιοποιήσουμε περισσότερο τα όσα μπορούμε να κάνουμε και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ και μπορεί να μας βοηθήσει για αυτά, διότι υπάρχουν... Ε, εδώ υπάρχουν εκεί ορισμένοι που λένε ε, easy boys που, και εδώ που εκπροσωπούν την Κομισιόν. Ίσως μπορούν να λάβουν το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ως πρόεδρος θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας τη γνώμη που θα υιοθετήσουμε από την Επιτροπή Ρέτζη να τονίσουμε την συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα δύο μέσα, την σημασία της, του μέσου πολιτικής, πολιτικής συνοχής και τις διαφορές βεβαίως. Έχουμε διαφορετικούς στόχους διαφορετικά κονδύλια, όπως είπατε, αλλά ταυτόχρονα θα, θα πρέπει να τονίσουμε την σημασία και τον ρόλο της πολιτικής της συνοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μέρος των σχολείων των συναδέλφων. Μήπως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να απαντήσω πολύ σύντομα σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ε, συμφωνούμε με τις απόψεις του συντάκτη και του κυρίου Τζέλερ όπως τα συνόψισε. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ποιος είναι ο, τελικός στόχος του επενδυτικού σχεδίου του Προέδρου Γιούνκερ. Ο στόχο είναι να ενισχύσουμε την ποιότητα των επενδύσεων ώστε να αρχίσει μια ροή επενδύσεων και η χρηματοδότηση είναι μόνο ένα από του τρει βραχίονες. Ε, το βασικό στοιχείο για τα μέσα χρηματοδότηση. Ε, ε, δεν έχουν καθοριστεί ακόμα, αλλά νομίζω ότι συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με αυτά τα οποία είπαν αρκετοί από τους ομιλητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ότι ένα, το κριτήριο, ένα κριτήριο είναι μεν οικονομική και τεχνική αξιοπιστία, αλλά ε, οι κατάλληλοι όροι είναι ένα βασικό... Ε, ε, ε στοιχείο του σχεδίου Juncker και δεν κανιβαλίζουμε όπως είπατε. Ένα από τους βασικούς στόχους είναι η κινητοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου και αυτό με οδηγεί στο επόμενο σημείο το οποίο αναφέρθηκε από αρκετούς ε, ομιλητές. Ε, πράγματι θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν είναι ένα νέο μέσο πολιτικής συνοχής, δεν υπάρχει κάποια ε, ως ε, διπλό ταμείο, είναι ένας τρόπος να ξεκινήσουν να εισραίουν επενδύσεις που στη συνέχεια σε δεύτερο βαθμό θα έχει και θετικές συνέπειες για τις περιφέρειες. Αλλά επειδή θέλουμε να έχουμε συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη επιλογή προγραμμάτων. Δεν υπάρχει τίποτα ε, αρνητικό ή θετικό σε σημείο διάκρισης, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει κάποια γεωγραφική προδιάθεση, αν θέλετε. Θεωρώ σε γενικέ γραμμέ ότι ελπίζουμε ότι οι θετικέ συνέπειε ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγών Επενδύσεων θα βοηθήσουν να έχουμε ε, επενδύσει σε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τις ε, τροπολογίες που υπευλήθησαν, δεν θα τις διατρέξω όλες μία προς μία ε, και του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Όσον αφορά τις εκθέσεις, σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν εκθέσεις και αξιολόγηση. Το τι απαιτείται ε, ελπίζω να δείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία σε σχέση με το άχθος αυτών που θα πρέπει να δηλώσουμε. Μπορεί να υπάρξει και μια αξιολόγηση που προβλέπεται και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ε, και να εξισορροπήσουμε συγγνώμη, το κόστος και τα ωφέλη σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει βεβαίως ε, και το θέμα της πράξης κατά εξουσιοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι βέβαιη ότι είναι απαραίτητη, ε, δεν είμαστε απόλυτα κατά, αλλά αν αυτό αποφασίσετε να ακολουθήσετε θα πρέπει να δούμε και από νομική σκοπιά αν είναι εφικτό να υπάρχει ε, ένα, ε, ε, μια τέτοια πράξη κατεξουσιοδότηση. Και με αυτό ολοκλήρωσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επενθυμίσω σε όλους την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 5 Μαρτίου, το γενέθλιο του κυρίου ε, και δεχτά όλα τα δώρα αλλά μόνο στα αγγλικά. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ε, έχουμε μάλλον δύο σημεία τα οποία είναι αλληλένδετα, τα σημεία 11 και 12. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Βίκτορ Μποστινάρου, ο οποίος ε, έχει πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του σήμερα. Ελπίζω όμως να έχει αρκετό χρόνο για να μας παρουσιάσει τις ε, γνωμοδοτήσεις του για τα δύο αυτά σημεία μαζί, διότι ε, έχουν σχέση μεταξύ τους. Το ένα είναι η τροποποίηση του κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρατόμα υπαρισμό 1311 του 2013 για τον καθορισμό του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 και το επόμενο σημείο είναι το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 2 του 2015 για τη μεταφορά πιστώσεων, επιμερισμένη διαχείριση, οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή, βιώσιμη ανάπτυξη, ασφάλεια και ηθαγένεια και η Ευρώπη στον κόσμο. Συντάκτης ο κύριος Ποστινάρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά γιατί έχω το σημειώσει μου στα αγγλικά και θα προσπαθήσω εδώ να εξηγήσω γιατί ακολουθούμε κάποιες από αυτές τις διαδικασίες, γιατί γίνονται τα πάντα μόνο στα αγγλικά και γιατί θα πρέπει να εγκριθούν αυτά το συντομότερο δυνατόν εν ευθέτω χρόνο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και κάποια αποτελέσματα. Οι δύο γνωμοδοτήσεις που σας παρουσιάζω σήμερα ε, αφορούν ε, την ε, μάλλον έχουν ως επί αρμόδια επιτροπή την Επιτροπή Προϋπολογισμών και μας ενδιαφέρουν τα επιχειρησιακά προγράμματα για τη νέα προγραμματική περίοδο. Θα σας παρουσιάσω τις δύο γνωμοδοτήσεις από κοινού, διότι ε, είναι αλληλένδετες. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαρθρωτικών Επενδύσεων, είχαμε μόνο 251 επιχειρησιακά προγράμματα, δηλαδή 43% του συνόλου που εγκρίθηκαν μέχρι το τέλος του 2014. 75 επιχειρησιακά προγράμματα, ήτι 17% του συνόλου, μεταφέρθηκαν βάσει του άρθρου 13 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, που σημαίνει ότι ήταν έτοιμα προς έγκριση στο τέλος του 2014 αλλά δεν υπήρξε δυνατότητα να εγκριθούν ε, εγκαίρως λόγω χρονικών περιορισμών. Επομένως αναβλήθηκε η έγκρισή τους για τις αρχές του 2015 και υπάρχει ακόμα δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι δεσμεύσεις του 2014. Για όλα τα υπόλοιπα ε, προγράμματα, τα 262 που απομένουν, που είναι το 45% του συνόλου, ούτε εγκρίθηκαν ούτε είναι ε, στη διαδικασία μεταφοράς και η μόνη διαδικασία που επιτρέπεται ώστε να μην χαθούν οι δεσμεύσει των κονδυλίων του 2014 είναι αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι την 1η Μαΐου βάσει του άρθρου 19 του, του κανονισμού για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δύο προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα να την ευχαριστήσω την Επιτροπή για το έργο και τη συνεργασία της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το γεγονός ότι πρέπει να εγκριθούν ε, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση. Λόγω χρονικών προδιορισμών όλες οι διαδικασίες των δύο θεμάτων γίνονται ε, στα αγγλικά μόνον και με πολύ σύντομες προθεσμίες. Επαναλαμβάνω πάρα πολύ σύντομες διορίες. Οι δύο γνωμοδοτήσεις έχουν δύο ε, διαφορετικές διαδικασίες όσον αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου ως συνήθως υπόκειται ε, στην ε, σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο διορθωτικού ε, προπολογισμού αριθμό 2 του 2015 που σχετίζεται με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού υπόκειται σε διαδικασία συναπόφησης. Όσον αφορά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί της οποίας έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο, είναι να μεταφερθεί σχεδόν ατόφιο το ποσό από το 2014 για τον τίτλο 1Β, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω της καθυστερημένης έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων το 2015. Αυτό σημαίνει ότι Ε, το βάρος θα το αναλάβουν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές το 2015, αλλά αυτό έγινε προκειμένου να διασφαλίσουμε ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών και υπ' αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα συμμετάσχει ενεργά και θα ε, βοηθήσει και στη διάρκεια του προγραμματισμού και στη ε, διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαναλάβει σήμερα τη δεσμευσή της να διαδραματίσει αυτό το ρόλο που σας ανέφερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να μεταφράσει αυτή τη δήλωση από τη θεωρία σε πράξη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να καθυστερήσει περαιτέρω με την έγκριση των υπόλοιπων προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή ε, εγκριθούν ε, και η αναθεώρηση του δημοσιονομικού ε, πλαισίου και το σχέδιο προπολογισμού. Το μόνο το οποίο δεν μεταφέρεται στο 2015 αφορά τις ε, ε, διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα διαμεθοριακά προγράμματα και το μέσο Ευρωπαϊκής Γειτονίας, ε, το EMI, το οποίο μεταφέρεται για το 2017. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται διαφορετική προσέγγιση είναι γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσει στην έγκριση του νομικού πλαισίου και κατά συνέπεια και στα προγράμματα και η περιπλοκότητα των προγραμμάτων ε, επίσης συνεισφέρει διότι περιλαμβάνουν τρεις φορεί κρατη κράτη-μέλη, υποψήφιες χώρες και γείτονες χώρες. Θεωρώ ότι για λόγους συνέπειας και προκειμένου να επιτρέπουμε και την ε, ταχύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων θα ήταν πιο λογικό να ακολουθήσουμε την ίδια λογική όπως και για τα υπόλοιπα ε, ποσά. Θα ήθελα να επισημάνω παρόλα αυτά ότι τα προγράμματα αυτά είχαν προβλεφθεί ήδη για το 2015 και το 2016 κάτι το οποίο ίσως θα μπορούσε να γίνει και θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ποσά. Εγώ βέβαια προτείνω να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας και διότι αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και τη χρήση των δεσμεύσεων του 2014 για τα επιχειρησιακά προγράμματα ε, δεν μπορούσαμε, που δεν μπορέσαμε να εγκρίνουμε το 2014 ε, βάσει της διαδικασίας μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή και η Επιτροπή ε, έχει ήδη τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου για να υποστηρίξει την πρόταση. Επομένω, πρέπει να ολοκληρώσουμε και εμεί τη διαδικασία μα και να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μα το συντημότερο δυνατόν. Και αυτό ε, θα ζητήσω και εγώ ε, σε όλους τους κοιόδης συζητητές και σε όλες τις πολιτικές ομάδες να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε αποτελεσματικά όπως έχουμε κάνει πολλέ άλλε φορέ. Το σχέδιο διορθωτικού υπολογισμού 2 του 2015 έχει άμεση σχέση με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, διότι μεταφράζει ουσιαστικά στην πράξη αυτό το οποίο αποφασίζεται στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου. Επομένως, τη μεταφορά σχεδόν όλων των τίτλων ε, του 1β ε, του 2014 που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο 2015. Αυτά έχουν συνολικά 16,5 δις ευρώ. Η άποψή μου ότι είναι ότι εδώ έχουμε κάτι αντίστοιχο με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου και δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Το μόνο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ε, επί τη ευκαιρία έθιξα για άλλη μια φορά το θέμα της καθυστέρησης των πληρωμών, οι οποίες ανέρχονται περίπου σε 25 δις ευρώ στο τέλος του 2014 για τα τρία κονδύλια. Γι' αυτό ακριβώς και στη γνωμοδότηση ζητώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ε, για την ε, κατάσταση ε, τι συνέπειες θα υπάρξουν κυρίως ε, ε, μεταξύ του 2017 και του 2018 όσον αφορά τις πληρωμές και επίσης το μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η καθυστέρηση των πληρωμών δεν θα επιδεινωθεί περαιτέρω. Το χρονοδιάγραμμα για τις δύο γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχο και να είναι το εξής έγκριση των δύο γνωμοδοτήσεων από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στην επόμενη συνεδρίαση τέλη Μαρτίου. Έγκριση στην Ολομέλεια τον Απρίλιο, στην πρώτη μικρή Ολομέλεια εδώ στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα επίσης να ε, κάνω έκκληση προς τους κοιόδης ε, εισηγητές και πάλι. Θα ήθελα να ζητήσω και την υπομονή τους και το γεγονός ότι μπορούν να εργαστούν σε πολύ στενά χρονικά προεριφέρεια. Γι' αυτό και ακριβώς ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι ο μόνος τρόπος να εγκριθούν αυτά εγκαίρως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια τα οποία απαιτούνται για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και επειδή γνωρίζω Γνωρίζω ότι οι τροπολογίες ε, δεν θα μπορέσουν να υποβληθούν. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι ε, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, σας ευγνωμονώ και ελπίζω να μπορέσουμε να εργαστούμε ώστε να τα εγκρίνουμε όπως έχει προβλεφθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να αναφέρω ότι ο κύριος Μποστινάρου με τον ίδιο σύντομο τρόπο και ο κύριο Φανιστερόη ετοίμασε την ε, έκθεση γιατί ε, αποφασίσαμε να γίνει αυτή η έκθεση στην ε, έκτακτη συνεδρία των συντονιστών στο Στρασβούργο. Σε εκείνη τη συνεδρίαση συζητήσαμε το πρόγραμμα για την προετοιμασία των εκθέσεων και προτιθέμεθα να υφετήσουμε αυτή την έκθεση στην επόμενη συνεδρία στις 26 Μαρτίου και γι' αυτό η Γραμματεία και εγώ ως Πρόεδρος προτείνω να δώσουμε μια προθεσμία για υποβολή τροπολογιών στα αγγλικά μόνο στην ίδια ε, περίφημη ημερομηνία της 5ης Μαρτίου. Αυτή είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών και αυτό ε, συμβαίνει για όλους τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν. Συνάδελφοι, ο λόγος σας κύριε Νοβάκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα υπάρχει μια γλώσσα εργασίας και έχουμε στενό χρονικό περιθώριο για να συνεργαστούμε σε αυτό το φάκελο. Αλλά πρώτα να πω ότι έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες ως προς το τι θα δοθεί από τον περιπολογισμό. δεν ήταν αυτό που περιμέναμε από το πολιτισμικό πλαίσιο και αν το Συμβούλιο θα δεχτεί να αυξήσει το όριο για τις ε, δεσμεύσεις. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και θα πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένα βήματα. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη θέση ως κοινοβούλιο για το πρώτο όριο των δεσμεύσεων προκύπτουν πολλά θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν για αυτήν την καθυστέρηση των ε, πληρωμών. Και τέλος, κάτι ακόμα σημαντικό. Είμαι βέβαιος ότι την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο να εργαστούμε, ώστε να έχουμε πιο ε, επικοδομητικές συζητήσεις, γιατί κάποια θέματα σίγουρα δεν θα ε, συζητηθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη εξαιτία του στενού χρονικού ε, πλαισίου. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Κυρία Ταμάτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Εξετάζοντας τα ποσά, ε, 300 επιχειρησιακά προγράμματα που είναι περίπου 47% των προγραμμάτων ε, για την κατανομή του δημοσιονομικού πλαισίου για να μην χάσουμε τους πόρους που έχουν διατεθεί το 2014 ανησυχώ ιδιαίτερα και την εκφράζω αυτή την ανησυχία. Ευπρόσδεκτη λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Θα ήθελα όμως καταρχάς να αναρωτηθούμε όσον αφορά την, το λόγο αυτής της καθυτέρησης. Όχι για να κατηγορήσουμε κάποιον οπωσδήποτε, αλλά για να δούμε ε, πώς μπορεί να μην επαναληφθεί αυτό στο μέλλον, στην επόμενη προγραμματική περίοδο και όσο το δυνατόν για να δώσουμε σωστέ πληροφορίε στου πολίτε και στους ψηφοφόρου μα. Όσον αφορά την περίπτωση τη Ιταλία, λίγο πολύ γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν, τα οποία λίγο πολύ είναι τα ίδια, όπω επεσήμενε και η ίδια η επίτροπο Κρέτσου, κυρίω για την ε, Νότια Ιταλία. Αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και το τεράστιο πρόβλημα των ε, ε, καθυστερήσεων των προϊλωμών στην πολιτική συνοχή και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λογοδοτήσει όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και όλο το σύστημα τη Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Ε, πρόκειται για 25 δις ευρώ τα οποία πρέπει να καταβληθούν στους ε, δικαιούχους όπως είπε και ο εισηγητής. Και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με το αίτημα του εισηγητή να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν πληροφορίες ε, ακριβής για το θέμα αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και από πολιτικής αλλά και από οικονομικής και κοινωνικής σκοπιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Βαν Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ε, συμμετοχή τους στη συζήτηση. Να επανέλθουμε πάνω σε αυτό, σε αυτή την μεταφορά κονδυλίων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι κάτι το εξαιρετικό. Τα δύο τελευταία σημεία, το 6 και το 7, σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015. Αυτό σημαίνει ότι ε, θα ληφθούν υπόψη. Εγώ νόμιζα ότι από πλευρά της Επιτροπής το θέμα μπορούσε να ρυθμιστεί. Είναι δύο θέματα τελείως διαφορετικά. Ε, υπάρχει το πρόβλημα των λογαριασμών που δεν έχουν πληρωθεί, των απλήρωτων και το πρόβλημα της ε, σύνδεσης των δύο. Thank you very much. Other wishes for contribution? No. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Κύριος Μποστινάρου, θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να πω στους ομιλητές ότι φαντάζομαι πως η Επιτροπή θα αντιδράσει για το αν αποδέχεται όλα αυτά και να γνωρίσετε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δέσμευση ότι η Επιτροπή θα εργαστεί ότι αυτά που μας υποσχέθηκαν θα εφαρμοστούν πλήρως παρέχοντας τη βοήθεια ε, στα κράτη-μέλη να ανακάψουν από αυτά τα προβλήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι οι καθυστερήσεις εντός των κρατών μελών για την προετοιμασία των επιχειρησιακών προγραμμάτων και επιπλέον καθυστερήσεις στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το πρόβλημα έγκυται σε δύο σημεία, όμως το πιο σημαντικό είναι να συνεργαστούμε και να διασφαλίσουμε ότι θα χειριστούμε το θέμα επαρκώς με την βοήθεια της Επιτροπής και με την κατάλληλη εφαρμογή, εκτέλεση εντός των κρατών μελών. Αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί το κοινοβούλιο μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα. Να εγκρίνει ή να απορρίψει τις δύο προτάσεις. Δεν θέλω καν να διανοηθώ την απόρριψη. Αν όμως εργαστούμε σωστά, θα πράξει το ίδιο και η Επιτροπή σε σχέση με τα προγράμματα αρρωγής προς τα κράτη-μέλη και από τα κράτη-μέλη στη συνέχεια και τις ε, περιφέρειες, στην εφαρμογή, εκτέλεση των προγραμμάτων. Με τις καθυστερήσεις είναι αληθές ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε τον τελευταίο χρόνο. Μειώθηκαν οι καθυστερήσεις και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και κυρίως για το Συμβούλιο και τα προβλήματα που προέκυψαν σε κράτη-μέλη είναι το εξή. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποδεχτούν ότι οι καθυστερήσει θα πρέπει να μετατραπούν σε πληρωμές και γι' αυτό χρειάζονται συνεισφορές οι οποίες πολλές φορές αμφισβητούνται. Βλέπετε λοιπόν το πρόβλημα είναι σε άλλα σημεία και σίγουρα όχι στο Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό το λόγο εμπιστεύομαι τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Επιτροπή και ο Επίτροπος και η Επίτροπος Ευρωπαϊκής Αναπτύξης κυρία Κρέτζου και το Κολέγιο των Επιτρόπων ότι θα κάνουν το μέγιστο δυνατό για να αποφύγουν τη συσσόρευση καθυστερήσεων γιατί αν συμβεί αυτό η μεταφορά των δεσμεύσεων για το 2015 συν αυτό που θα πρέπει να μεταφερθούν για το 2017 τότε θα ε, προκύψει ένα τεράστιο άχθος που δεν θα είναι εφικτό να ε, είναι πληρωτέο. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει το χέρι μας για να το αποτρέψουμε. Δεν θεωρώ επίσης ότι πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί και να κατηγορούμε την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς πρέπει να λάβουμε υπόψη ποιοι είναι οι λόγοι για την καθυστέρηση υιοθέτηση έγκρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων. Όταν 262 πρόγραμμα, ε, επιχειρησιακά προγράμματα δεν έχουν εγκριθεί, τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα. Συν 75 επιχειρησιακά προγράμματα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη και να δούμε κατά πόσο είναι ικανές οι τοπικές αρχές και οι κυβερνήσεις και κατά πόσο πληρώνουν τις ευθύνε τους για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η συζήτηση που θα πρέπει να συνεχίσει στον ε, διεθνικό ε, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι όμως θέλω να σας ευχαριστήσω για τις συνεισφορές σας και για την αποδοχή αυτής της διαδικασίας γιατί πραγματικά είναι το μόνο που μπορούμε να πράξουμε ε, δεδομένων των χρονικών περιορισμών. εμπιστεύομαι τη βούληση και την δημότητα αυτής της διακεκριμένης επιτροπής ε, ε, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν. 5 Μαρτίου δεν είναι τα γενέθλιά μου, αλλά θα ήθελα και εγώ θα δεχτώ συμβολικό δώρο για αυτή την ημερομηνία στα αγγλικά όμως παρακαλώ. Ευχαριστώ και επαναλαμβάνω η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών είναι η 5η Μαρτίου 12 το μεσημέρι και μόνο στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποστινάρου. Αναφέραμε πολλέ φορέ στην Επιτροπή, αλλά δεν έχουμε δώσει ακόμα το λόγο στου εκπροσώπου τη Επιτροπή. Σα δίνω λοιπόν το λόγο για να αντιδράσετε στα σχόλια που έχουν γίνει. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ ε, στον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να τονίσω ότι το θέμα αυτό είναι πήγον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η αναθεώρηση του πολιωτούς δημοσιονομικού προγράμματος και του σχεδίου προϋπολογισμού να υιοθετηθούν την 1η Μαΐου ούτω ώστε να μην καθυστερήσει περαιτέρω ε, η υιοθέτηση των προγραμμάτων 2014-2020. Έχουμε ε, στις 13 ε, Φεβρουαρίου την ε, συμφωνία στην Κορεπέρ που υιοθετήθηκε μία εβδομάδα μετά τυπικά από το ΕΚΟΦΗΝ. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη όπως λέχθηκε για να την έχουμε στην Ολομέλεια του Απριλίου, ούτως ώστε το Συμβούλιο να μπορεί την 1η Μαΐου να υιοθετήσει την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού ε, πλαισίου. Είχαμε δύο δηλώσεις, δύο ανακοινώσεις που καλύπτουν τις διάφορες ε, επιφυλάξεις ε, των αντιπροσωπιών και που μπόρεσαν να οδηγήσουν σε καλή πολιτική συμφωνία. Η πρώτη δήλωση εστιάζεται στην επίπτωση των μεταφορών των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων ούτω ώστε να διαβεβαιώσουμε τα κράτη-μέλη ότι το reprofiling δεν απαιτεί αλλαγές όσον αφορά ε, τις πληρωμές. Το, η δεύτερη που είναι πάρα πολύ σημαντική και αναφέρθηκε από μέλη της Επιτροπής είναι ότι η Επιτροπή ε, δεν θα αφιστεί καμιά προσπάθεια ούτως ώστε τα προγράμματα να υιοθετηθούν το συντομότερο δυνατόν και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα παράσχουμε την απαιτούμενη βοήθεια στα κράτη-μέλη ούτως ώστε τα κονδύλια τα οποία μεταφέρθηκαν με αυτήν την άσκηση θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μην χαθούν κονδύλια σχετικά με την καθυστέρηση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε ήδη στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαδικασίας για τον προϋπολογισμό 2015 και το Δεκέμβριο 2014 κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε μια κοινή δήλωση περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό 2015 σύμφωνα με την οποία συμφωνήθηκε ότι το πρόγραμμα πληρωμών για τις καθυστερήσεις πληρωμών για την προηγούμενη περίοδο 2007-2013 θα εγκριθεί από τις δημοσιονομικές αρχές πριν από την έναρξη της επόμενης διαδικασίας ε, της δημοσιονομικής. Είναι σημαντικό όταν μιλάμε για καθυστέρηση υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Υπάρχει μια κανονική καθυστέρηση και υπάρχει μια εξαιρετική έκτακτη ε, καθυστέρηση. Ε, στο τέλος του έτους αναφέρεται ε, σε αιτήματα τα οποία δεχτήκαμε αργά κατά τη διάρκεια του έτους σε διεκδικήσεις, αλλά έχουμε και καθυστερήσεις έκτακτες που υπάρχουν λόγω ελλείψεως πιστώσεων, διαθεσίμων πιστώσεων. Και είναι αληθές ότι αυτές οι καθυστερήσεις ε, δεν είναι σε τρέχον επίπεδο και αυτό το επίπεδο ε, δεν είναι βιώσιμο για μας. Γι' αυτό εργαζόμαστε τώρα για την προετοιμασία του προγράμματος ε, πληρωμών και στις επόμενες εβδομάδες η Κομισιό θα συμμετάσχουν σε διάλογο με τις ε, δύο, τα δύο σώματα ε, της ε, δημοσιονομικής αρχής για τα μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν ούτως ώστε το τέλος του έτους 2016 να έχει μειωθεί σημαντικά αυτή η καθυστέρηση. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα αυτό θα πρέπει να γίνει πρωτού αρχίσουμε τις συζητήσεις για την επόμενη δημοσιονομική διαδικασία. Γι' αυτό η Κομισιό έχει θα συμμετάσχει σε αυτό το διάλογο μαζί σας ε, σύντομα και θα παρουσιάσουμε διάφορα μοντέλα και διάφορες δυνατότητες για να μειωθεί αυτή η καθυστέρηση. Η συσσωρευμένη καθυστέρηση. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σε ένα τελικό θέμα είναι το reprofiling, η εκπόνηση ενός ε, νέου προφίλ ε, με τα διάφορα στοιχεία, είπα και είναι και προτείνουμε έναν επαναπρογραμματισμό για το μέχρι το έτος 2017 και θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί προτείνουμε αυτό το νέο προφίλ. Πρώτον, είναι σαφές ότι η εκπόνηση των προγραμμάτων αυτών παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από τα προγράμματα των κρατών μελών, διότι πρέπει να συνεργαστούμε με εταίρους από υποψήφιες χώρες και χώρες της, του προγράμματος γειτονία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι τη νομική βάση για την, το ΙΠΑ και το ΙΕΝΑ, για τα δύο αυτά μέσα, υιοθετήθηκαν αργότερα ε, θυμάστε ότι η νομική βάση μας υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο 2013, ενώ η νομική βάση για το ΙΠΑ και η ΕΝΑΗ τον Μάρτιο 2014 και αυτό εξηγεί την καθυστέρηση. Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι παρόμοια προσέγγιση προτάθηκε στο έτος 2008 με την προηγούμενη περίοδο όπου ε, τα ποσά ε, μεταφέρθηκαν τα κονδύλια σε επόμενα έτη. Αυτό εξηγεί την διαφορετική προσέγγιση ως προς τα προγράμματα αυτά. Και πάλι ευχαριστώ για την προσοχή σας, για την υποστήριξή σας σε αυτό το σημαντικό πολιτικό φάκελο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρα. Έχουμε κλείσει την εργασία μας για αυτά τα δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης. Σας Υπενθυμίζω ότι αποφασίσαμε να, να προσθέσουμε ένα πρόσθετο σημείο σχετικά με τις, τους κανονισμούς της Κομισιόν μετά τον Φεβριάριο 2015 που να ε, το, το κανονισμό 480 να θεωρούν το 2014 σε σχέση με στον κανονισμό 508 του 2013 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Κομισιό υιοθέτησε αυτές τις κατεξοδότηση πράξεις ε, προσπαθώντας να ε, ε, αναθεωρήσει τον κανονισμό για την θάλασσα και την αλληλεία και ε, μια προηγούμενη, κανονισμό προηγούμενος κανονισμός έπρεπε να λάβει υπόψη την θέση σε ισχύ του σχετικού Ταμείου Αλληλείας, του κανονισμού του Ταμείου και των διατάξεων. Πρόκειται για μια τεχνική πρόταση που κοινοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο σε όλες τις γλώσσες στις 13 Φεβρουαρίου και μετά σας κοινοποιήθηκε με email το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει το σχέδιο ψηφίσματος το συντομότερο δυνατόν με βάση τις αιτίες για τις οποίες αντιτίθεται ε, κανόνας 105 σε δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής της περίοδου για αντιρρήσεις αν ε, η Επιτροπή δεν ε, λάβει μέτρα ε, θα ε, θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Τώρα δίνω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιό ε, για να εξηγήσει τον στόχο της κατεξιοδότηση πράξης Αλεξ Παυριτσάνη. Δεν ξέρω αν πρόφερα καλά το όνομά σας, σας δίνω τον λόγο. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Υπενθυμίσατε πολύ καλά λίγο το ιστορικό. Έχουμε έρθει λοιπόν για τροποποίηση ε, τεχνικής φύσεως Πρόκειται για τον κανονισμό 470 του Μαρτίου του 2014. Εγκρίθηκε το Μάρτιο γιατί δεν μπορούσαμε να περιμένουμε την έγκριση του κανονισμού για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και πρέπει να κάνουμε κάποια μελλοντική αναφορά στον κανονισμό ε, αυτό. Αυτή τη στιγμή εγκρίθηκε ο κανονισμός το Μάιο του 2014 μπορούσαμε να αλλάξουμε και να αντικαταστήσουμε τις προκαταρκτικές παραπομπές ε, του κανονισμού για την ε, καταξουσιοδότηση πράξη με τις σωστές αναφορές ε, για τον κανονισμό για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επιπλέον διορθώσαμε και το παράρτημα 3. Το παράρτημα 3 είναι ο κατάλογος των δεδομένων που θα πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε ψηφιοποιημένη μορφή. Πρόκειται λοιπόν για αρκετά τεχνικό σημείο και υπήρχε και κάποια αναφορά στο δημοσιονομικό πλαίσιο για τις συμπράξεις ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Ε, αυτά ε, εξηγήθηκαν στην ομάδα για τις εκτελεστικές και πράξη και τη πράξη κατά εξουσιοδότηση, παρουσία και πυρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 και το επόμενο βήμα πλέον, εφόσον κοινοποιήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το, το Φεβρουάριο και όπως είπατε και εσείς, το επόμενο βήμα είναι... Ε, εντός αυτών των δύο μηνών, εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις, να τεθεί σε ισχύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ωραία, σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος από τα μέλη της Επιτροπής ε, Ρέτζι που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ε, όχι. Προτείνω λοιπόν είναι η Επιτροπή να μην ζητήσει παράταση για το διάστημα των δύο μηνών που επιτρέπεται για ένσταση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και η πρότασή μου είναι να θέσουμε μια προθεσμία 12 το μεσημέρι, 3η 3 Μαρτίου, για, αποσταλή, για να αποσταλούν στη Γραμματεία ε, οποιοδήποτε κείμενο το οποίο ε, έχει αντιρρήσεις για το συγκεκριμένο κείμενο. Ε, συμφωνείτε? Ναι, συμφωνούν λίγο πολύ τα μέλη. Σας ευχαριστώ. Αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. The next point is any Το επόμενο σημείο είναι τα διάφορα. Υπάρχει κάτι από τα διάφορα. Όχι. Δεν έχουμε λοιπόν τίποτα στα διάφορα. Να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 26 ε, Μαρτίου, ημέρα 5η, 9 με 12.30 και 3 με 6.30 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για την υποστήριξή τους ε, στη διάρκεια της συνεδρίασης μας πέρα τη συνεδρίαση, αλλά να ζητήσω από τους συντονιστές να παραμείνουν για συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών των συντονιστών. Ευχαριστώ.